Bene, Τροποποίηση του κανονισμού ΕΚ αριθμός 1698-2005 του Συμβουλίου. Συνάδελφοι, σημείο 6 στη 8, συγγνώμη, στην ημερήσια διάταξη. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στην περασμένη μας συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, εκφράστηκαν ανησυχίες επειδή αυξήθηκαν οι πληρωμές για τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 και 2012. Και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το συνολικό χαρτοφυλάκιο που διατίθεται για τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου στα διάφορα Αφού εξετάσαμε την πρόταση κατά λεπτός, φαίνεται ότι ο κίνδυνος αυτός δεν είναι τόσο σοβαρός. Σοβαρότερος είναι εκείνος το να χαθούν συνολικά οι εγγεγραμμένοι στον προπολογισμό, οι εγγεγραμμένοι στον προπολογισμό ευρωπαϊκής πληρωμές, λόγω της έλλειψης κρατικών κονδυλίων. Γι' αυτό λοιπόν πρότεινα και προκειμένου να στηριχθούν οι οικονομίες της Υπέθρου και γενικότερα η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επιταχύνουμε την νομοθετική διαδικασία ώστε να αρχίσει να ισχύει πριν το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, πριν το τέλος του 2011. Για το σκοπό αυτό υπέβαλα την έκθεση αυτή χωρίς όμως ε, νομοθετικές τροπολογίες στην πρόταση. Παρόλα αυτά, συνάδελφοι, αυτή την εβδομάδα μάθαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Προβλήματα γιατί το Συμβούλιο θέλει να εξέβρει οριζόντια λύση και για τα υπόλοιπα διαφορετικά ταμεία. Έτσι, επειδή η έγκριση στο Συμβούλιο έχει μπλοκαριστεί προς στιγμή, λόγω αυτών των εξελίξεων, το ζήτημα αυτό μπορούμε να το δούμε κατά τον ιωθώτα τρόπο, δηλαδή ορίζοντας προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 26 Οκτωβρίου, ενώ θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. Θα θέλαμε να είμαστε ταχύτεροι, αλλά δεδομένου του μπλοκαρίσματος στο Συμβούλιο, θα κάνουμε ό,τι θα κάναμε ούτως ή άλλως. Ο κύριος Άγνιο έχει ζητήσει το λόγο. Υπάρχουν εδώ και εκπρόσωποι της Επιτροπής, ο Διευθυντής Μαρίνο είναι εδώ. Εφόσον υπάρξουν λοιπόν ερωτήσεις ή απορίες από τους συναδέλφους, θα μπορούμε να έχουμε απαντήσεις. Κύριε Ανιώ, Πρόεδρε, αυτή η αναθεώρηση του εξαετούς κανονισμού σημαίνει ότι 150 εκατομμύρια ευρώ για την φετινή χρονιά, 560 μάλλον εκατομμύρια ευρώ, 90 φέτος και 70 του χρόνου, θα εκταμιευθούν. Πώς θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια. Το μόνο που λέγεται από την πρόταση της Επιτροπής είναι ότι θα αναρωθεί ανάγκη για πρόσθετες πληρωμές και εκταμιεύσεις και εφόσον χρειαστεί, θα προτεθούν σχετικές δράσεις στην ε, αρχή προπολογισμού. Σε απλά αγγλικά, αυτό λέει ότι θα πάρουμε τα κονδύλια αυτά, ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα το προσέξει και θα κάνουμε τα πράγματα έτσι ώστε να σα πείσουμε να προσβλέψετε πρόσθετα κονδύλια σε δύο χρόνια. Το σχόλιο στο επεξηγηματικό σημείωμα λέει και παραθέτω εδώ ότι η πρόταση τη Επιτροπή δεν προβλέπει ε, πρόσθετε ε, οικοδαμιεύσει για το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα απόλυτο και ξεκάθαρο ψέμα. Μα, Κύριε Ανιώ, θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή Μαρίνο για να μπορέσει να σας καθησυχάσει σε σχέση με αυτήν την απειλή που διαβλέπετε. Αλλά να καθησυχάσω τους συναδέλφους. Η τροποποίηση του κανονισμού για την οποία συζητάμε δεν αλλάζει καθόλου τον κοινοτικό προπολογισμό, δεν τον επηρεάζει. Επηρεάζει την συμμετοχή μεταξύ, που μοιράζεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 100 μελών για τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Υπό το πρίσμα λοιπόν του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, του γενικότερου προπολογισμού δεν υπάρχει καμία ε, συνέπεια. Απλώ ευελιξία στο εσωτερικό των, προγραμμάτων ανάπτυξη τη υπαίθρου. Τα κράτη-μέλη που έχουν δυσχέρειε να εντοπίσουν εθνικά κονδύλια, να εξεύρουν εθνικά κονδύλια, επιχρωτικά σήμερα για τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου, θα μπορούν να το κάνουν και με μια ποσόστοση χρηματοδότηση πιο χαμηλή. Στι συγκεκριμένε χώρε θέλουμε να μην υπάρξει μείωση των μέτρων για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Οπότε δεν υπάρχει καμία επίδραση για την προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. η Τροποποίηση του κανονισμού δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Όμω ο κύριο Μαρίνο θα μα τα εξηγήσει καλύτερα. Ή κυρία Μαρίνο μάλλον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό που είπατε είναι απολύτω ορθό. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με όσα προβλέπει ο προπολογισμό ήδη. Ιδίως για τις δαπάνες. Τώρα, οι δαπάνες πληρωμών. Οι πιστώσεις πληρωμών. Μιλήσατε για 470 εκατομμύρια επιπλέον για τις πληρωμές για το 2012. Ο αριθμός όμως αυτός θα πρέπει να εξεταστεί. Μιλάμε για 14 δις περίπου δαπανών, ε, πιστώσεις πληρωμών για το 2012. Είναι σχεδόν μηδαμινό. Ακόμη και από την άποψη των δαπανών, των πιστώσεων πληρωμών είναι ελάχιστο το ποσοστό αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διευκρίνηση. Ας υποθέσουμε ότι ένας γεωργός προτίθεται να κάνει μια επένδυση 100.000 ευρώ. Ας υποθέσουμε επίσης ότι το, η ελληνική η ισπανική αρχή λέει ότι η συγχρηματοδότηση είναι της τάξης του 70% και επομένως 30% βαραίνουν τον ίδιο τον Γιώργο. Άρα στην αναλογία αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Τα 70% του δημοσίου χρήματος η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή θα έχει 20% η Ελλάδα, 80% η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως τώρα το 80% του ευρωπαϊκού τμήματος μπορεί να αναχθεί στα 90 έτσι ώστε η Ελλάδα να κληθεί να δώσει μονάχα 10% του 70%. Άρα ο Γεωργός θα, θα πληρώσει τα 30%, θα καταβάλει τα 30%, η επιδότηση θα είναι της τάξης του 70% αλλά μέσα στην ίδια τη δημόσια επιδότηση αλλάζει η αναλογία των τμήματων Ευρώπης και Ελλάδος. Ναι, έτσι είναι, αλλά θα προτιμούσα να το ακούσουμε από τη Διευθύντρια Μαρίνο. Ναι, σωστό. Η αναλογία που καλύπτεται από την Ευρώπη και στο παράδειγμα, αν προκειμένου η Ελλάδα, αλλάζει. Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τη συνεισφορά των ίδιων των γεωργών. Απλώ, ακριβώ επειδή αυξάνεται η αναλογία χρηματοδότηση τη Ευρώπη, το μέτρο θα, μπορούσε να, μπορεί τελικά να εφαρμοστεί. Ιδάλω, τελικά να μην ήταν σε θέση να ισχύσει. Διότι δεν υπάρχει αρκετή εθνική συγχρηματοδότηση. Πολύ ωραία. Νομίζω οι διευκρινήσει τη Διευθύντρια Μαρίνο ήταν αρκετέ θα υπήρχε στρέβλωση του ανταγωνισμού εάν υπήρχε διαφορετική συμμετοχή των γεωργών στα κράτη-μέλη. Παραμένει ίδια, ίδια παντού η συμμετοχή. Αυτό που αλλάζει είναι η συμμετοχή δημόσια, δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών, η αναλογία μεταξύ του. Και αυτό για να επιτρέψουμε στα κράτη που έχουν οικονομικέ δυσχέρειε να μην δαπανίσουν του πόρου του, επειδή ακριβώ δεν μπορούν να εντοπίσουν το ανάλογο εθνικό κονδύλι. Βάσει λοιπόν των πρόσφατων εξελίξεων, μπορούμε μάλλον να το ξανασυζητήσουμε το θέμα, εφόσον αναβλήθηκε στις 26 Οκτωβρίου η εξέταση και εφόσον το Συμβούλιο θέλει να συζητήσει και τα υπόλοιπα διαφορετικά ταμεία. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα έλεγα να περάσουμε απευθείας στο επόμενο σημείο, το σημείο 9. Υγεία των μελισσών και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα. Εισηγητής ο κύριος Ταμπάτζη τον οποίο βλέπω στη θέση του και τον χαιρετώ. Συνάδελφοι, θα δούμε τώρα την έκθεση πρωτοβουλία του κυρίου Ταμπάτζη για το θέμα των προκλήσεων στον τομέα των μέλισσοκομικών. Έχουν υποβληθεί 220 τροπολογίε. Και για αυτέ βρέθηκαν 18 συμβαστικέ τροπολογίε, χάρη στη συνεργασία του, του και των υπολείπων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ψηφοφορία. Άριστο το, η προσπάθειά σου, και εσένα Τσάμπα και των σχεδόν εισηγητών. Θα ψηφίσουμε λοιπόν για 10 παραγράφους ενώ οι υπόλοιπε 46 καλύπτονται από την έκθεση. Συνάδελφε Τσάμπα θέλετε την, ε, το λόγο πριν την έκθεση. δάλλως θα ψηφίσουμε αμέσως. Παρακαλώ ετοιμάστε τις κάρτες σας. Κύριε Ταμπάτζη. Like Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους, τους κοιόδης ηγητές, την Πιελότσιλ, του βοηθό μου, τον Χάραλτ, τον Κρίστοφερ, τους συναδέλφους από το ΕΛΚ, την Ελλάδα, τη Μάλτα για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νταντάν, την κυρία Λούλινγκ, σε όλους τις θερμές ευχαριστίες. Ωραία, ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε στην ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι στο έτοιμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 48. 48. Εψήφισαν άπαντες. 48. 48. Πέρας. Εγκρίνεται. Ναι. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 4. Συμβεβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβεβαστική τροπολογία 4. Εψήφισαν άπαντε πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Μορφάει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 59. 60. Τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 60. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 61. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Σιλβέστρης. Άρχεται η ψηφοφορία για την 72. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ξανά για την τροπολογία 72 Σιλβέστρης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Καλά τα πήγαμε. Με μία ψήφο διαφορά πέρασε. Εγκρίνεται. 73. Τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία για την 73. 73. Πέρας. Η 73 εγκρίνεται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Τροπολογία 74. Άρχεται η ψηφοφορία για την 74. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχω... 77. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 77. Πέρας. Απορρίπτεται. Πηδήξαμε την 75 Ρούμπιξ. Την ξεχάσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 75 Ρούμπιξ. Πέρας. Η 75 απορρίπτεται, θα έλεγα. 78. Άρχεται η ψηφοφορία για την 78. Απορρίπτεται. 79. Άρχεται η ψηφοφορία για την 79. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 80. Τροπολογία 80. Δεν ψήφισαν άπαντε. Η τροπολογία 80 απορρίπτεται, μου φαίνεται. Απορρίπτεται. 81. Τροπολογία 81. Άρχεται η ψηφοφορία για την 81. Λούλιν και άλλοι. Πέρας. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. 82. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 82. 8-2. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. Ναι, απορρίπτεται. 83. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 83. Εψήφισαν άπαντε για την 83. Απορρίπτεται. 84. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 84. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. Άρχεται η ψηφοφορία για τον 85. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 86. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 86. Ψηφίζουμε για την 86. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος 18, ένβη 18, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν εγκρίνεται. Νόπασερα. Απορρίπτεται. Το περιβάλλον δεν τα κατάφερε. 87. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 87 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. 88. Τροπολογία 88. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 88. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Η συμβαστική 6 εγκρίνεται. 95. Τροπολογία 95. Ashworth. Άρχεται η ψηφοφορία για την 95. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 7. Τροπολογία 104. 104. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 105. 105. Πέρας. Η 105 εγκρίνεται. Η 105 απορρίπτεται, με συγχωρείτε. 106. 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 107. Άρχεται η ψηφοφορία για τον 107. Πέρας. Εγκρίνεται. 109. Άρχεται η ψηφοφορία για την 109. 109 πέρας. Εγκρίνεται. 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 110 εγκρίνεται. 111. Πάξας. 111 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 111 μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. 112. Άρχεται η ψηφοφορία για την 112. 112. Πέρας. Απορρίπτεται. 113. Ψηφίζουμε για την 113. Εψήφισαν άπαντες στην 113. Πέρας. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Εγκρίθηκε. Συμβεβαστική πρόταση 8. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η συμβαστική 8 εγκρίνεται. 117. Άρχεται η ψηφοφορία για την 117. Πέρας. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. ΕΝΒΙ 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Να περάσει αυτή. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε τώρα την συμβιβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβιβαστική 9. Πέρας. Εγκρίνεται. 121. Άρχεται η ψηφοφορία για την 121. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Η 121 απορρίπτεται. 122. Άρχεται η ψηφοφορία για την 122. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 της Επιτροπής Περιβάλλοντος πέρας. Απορρίπτεται μου φαίνεται. «123. Άρχεται η ψηφοφορία για την 123. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 10. Πέρας. Εγκρίνεται. 132. Άρχεται η ψηφοφορία για την 132. Πέρας. Νομίζω εγκρίνεται. NV9. Τροπολογία για 9 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πέρας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμμεβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμμεβαστική 11. Πέρας. Εγκρίνεται. 139. Λαβία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 139. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε τον Λαβία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβεβαστική 12. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 152. 152. Πέρας. Οι 152 μάλλον εγκρίνεται. NV10. Περιβάλλον 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 13. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. nv 36. Άρχεται η ψηφοφορία. NV36. Εψήφισαν άπαντε. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Πέρα. Η συμβαστική 14 εγκρίνεται. 168. Άρχεται η ψηφοφορία για την 168. Πέρας. Για την 168. Εγκρίνεται. Εκατόν Πέρας. Η 162 εγκρίνεται. 164. 174 μάλλον. Άσπορθ. Πέρας. Η 174 μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. 175. 175. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 175 απορρίπτεται. Envy. NV39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η NV39 απορρίπτεται. NV40. Άρχεται η ψηφοφορία για την NV40. Απορρίπτεται. NV41 τέλος. Άρχεται η ψηφοφορία για την NV41. Τα ίδια μου φαίνεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 15. Εψήφισαν απαντές. Εγκρίνεται. 179 Λαβία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 179. 179. Κλείνει. Απορρίφθηκε. Όχι εξαιτία του Πρόεδρου. 180. Ψηφίζουμε την 180. Άρχεται ε, ψηφοφορία για την 180. Πέρας. Απορρίπτεται. 182. Νταντέν. Υπάρχει όμως και προφορική τροπολογία από το Μισελ. Μισό το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω καταθέσει τροπολογία, διότι όπως έχει συνταχθεί το κείμενο, τεχνικός δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενιαία τροπολογία η συμβαστική για αυτή την παράγραφο. Θέλουμε να υπάρχουν τιμέ αναφορά. Ζητούμε λοιπόν για τα κτηνιατρικά προϊόντα που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ένα όριο τιμή αναφορά για τι παρεμβάσει ένα όριο το οποίο να ορίζεται σε 10 ppb για όλα τα εργαστήρια της Ένωσης δεδομένων των αναλύσεων που ε, χρησιμοποιούνται σε όλα τα κάτι μέλη. Ευχαριστούμε, Μισελ, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από συνάδελφο, να ψηφίσουμε για την τροπολογία με την προφορική διόρθωση. Ψηφίζουμε, λοιπόν, τροπολογία 182 με αυτή την διευκρίνηση. Πέρας. Μισελ μας έπεισες όλους. Εγκρίνεται. Όχι όλους, τέλος πάντων. Δεν συμφωνούν κι όλοι. 184. Άρχεται η ψηφοφορία για την 184. 184. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 185. Άρχεται η ψηφοφορία για την 185. Πέρας. Εγκρίνεται. Τη μια έτσι την άλλη αλλιώ. Τι να πω κι εγώ. Ποιο μου λέει τι έγινε, εσύ εκείνο. Τροπολογία 16. Συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία για την 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 190. Ψηφίζουμε για την 190. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 191. Ε, άρχεται η ψηφοφορία για την 191. Πέρας. Εγκρίνεται. 193. Άρχεται η ψηφοφορία για την 193. 193. Πέρας. Η 193 εγκρίνεται. 194. Άρχεται η ψηφοφορία για την 194. 194 πέρα. 194 απορρίφθηκε. 195. Άρχεται η ψηφοφορία για την 195. Η 195 ψηφίζεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 17. Πέρας. Η συμβαστική 17 εγκρίθηκε. Και τώρα 201. Άρχεται η ψηφοφορία για την 201. πέρα. Η 201 μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Ναι. 202. Γκαρσία Περέ. 202. Πέρας. Εγκρίθηκε. Νεντέλτσεβα 203. Άρχεται η ψηφοφορία για την 203. Πέρας. 203. Εγκρίνεται. 205. Νεντέλτσεβα. Ναι, Άρχεται η ψηφοφορία. 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 205 εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 18. Πέρα. Εγκρίνεται. 214. Νταντέν. 214. Άρχεται η ψηφοφορία. 2-1-4. Αυτή τη φορά ο Ζωζέ ψηφίζει το ίδιο με τον Ταντέν. 2-1-4 4 περα Ευρία πλειοψηφία. 215. Άρχεται η ψηφοφορία 2-1-5. 2-1-5 5 περα Εγκρίνεται. Ναι. Μου το επιβεβαιώνουν. Ψηφίζουμε για το 218. 218. Άρχεται η ψηφοφορία για την 218. Πέρας. 218 εγκρίνεται. 219. Κοσμάρεκ. 219, άρχεται η ψηφοφορία, 219, πέρας. Η 219 απορρίπτεται. Και τώρα, 220. Ψηφίζουμε για την 220. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε κάποιες αιτιολογικές αναφορές. Πρώτη. Ένα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται, νομίζω. Δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρόμοια αποτελέσματα. Εγκρίνεται. Τρία. Χάρκιν. Την τρίτη, αιτιολογική αναφορά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Συμβιβαστική τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αιτιολογική σκέψη εδώ. Εγκρίνεται. 8. Ψηφίζουμε την 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική την ε, τροπολογία 1. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 10. Πέρας. Εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. 12. Ταραμπέλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν μπορώ να καταψηφίσω τον Ταραμπέλα. 12. Πέρα. Απορρίπτεται. 13. Άρχεται η ψηφοφορία για την 13. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. Πέρα, Απορρίπτεται. 15. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Πέρα. Παρόμοια αποτελέσματα απορρίπτεται. 16. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη C. 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Εντέλτσεβα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 11. Πέρα. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία για την ατολική σκέψη. 17. Πέρα, πέρα. Απορρίπτεται. 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Όχι. Α, τώρα. Πέρα. Εγκρίνεται. 19. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 2. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογιατρία. Η συμβαστική τριά εγκρίνεται. 40. Δαντέν. Πέρα τη ψηφοφορία για την 40. Μισελ, αυτή τη φορά φοβάμαι ότι δεν πέρασε. Κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 39. Άρχεται η ψηφοφορία για την 39. Πέρας. Θα έλεγα ότι εγκρίθηκε. 41. Άρχεται η ψηφοφορία για την 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Άνοιξε. Ωραία. Τώρα άνοιξε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 42. 43. Με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 43. Πέρας. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Άρχεται η ψηφοφορία για την 47. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα τα ψηφίσματα. Α, φινία, φινάλε. Τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν απαντές. Ωραία. Το ψήφισμα λοιπόν, όπως έψηφισατε, 32 ψήφους υπέρ, μία κατά, τρεις αποχές. Με αυτές τις ψήφους εγκρίνεται. Συγχαρητήρια τα Ταμπάτζη. E Περνάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη. Το έχετε όλοι μπροστά σας ή θέλετε ένα break χάρτη πορεία για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρωπούχων εκπομπών το 2050. Εισηγητή, ο κύριο Μπέλα Γκλατφέλντερ. Συνάδελφοι, όπω τα γνωρίζετε, στι 19 Σεπτεμβρίου χρειάστηκε να αναβάλουμε την ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση του κυρίου Γκλατφέλντερ. Υποβλήθηκαν 68 τροπολογίες για το σχέδιο έκθεσης και ο εισηγητή μαζί με του Κεώδε ετοιμάσαν μία σειρά από συμβαστικέ αστροπολογίε για να διευκολυνθεί η ψηφοφορία. Κύριε Γκλάτε Φέλντερ, θέλετε την, ε, το λόγο. Ωραία, τότε ψηφίζουμε ευθύ αμέσω. Ξεκινάμε γρήγορα. Γρήγορα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία με τη συμβαστική 1. Πέρα τη ψηφοφορία. Η συμβαστική 1 εγκρίνεται. Adesso votiamo l'emendamento 7. Τροπολογία 7. George Lyon και Λένα Τροπολογία 7. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 8. Άρχεται η ψηφοφορία για την 8. Ξεκίνα. Άρχεται ε, έναρξη, πέρας. Απορρίπτεται. 9. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απροβάται. Γκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 2. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Τροπολογία 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Τροπολογία 17. Πέρας της ψηφοφορίας για την τροπολογία 17. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 3. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Αντσίλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Τροπολογία 25. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Όχι. 29. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται μάλλον. Ναι, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 29. Ξεκίνα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Πέρας. Απορρίπτεται μάλλον. 28. Τροπολογία 28. 28. Πέρας. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Ναι. 31. Άρχεται η ψηφοφορία για την 31. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας για την 31. Ισοπαλία. Απορρίπτεται. 32. Άρχεται η ψηφορία για την 32. Πέρας. Παρά τη στήριξη, βλέπει Τζοβάνι. Εγκρίθηκε. Ε, τροπολογία 4, συμβαστική 4. Εψήφισαν άπαντες για την 4, πέρας. Εγκρίνεται. 37. Τροπολογία 37. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 38 πρώτο τμήμα. 38 πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 38 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 39. Ψηφίζουμε για την 39. Πέρα. Απορρίπτεται. 40. Άρχεται η ψηφοφορία για την 40. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. 41. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. 42. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 43. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία για την 44. Πέρας. Η 44 εγκρίνεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία για την 45. Ίδια αποτελέσματα. Εγκρίνεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία για την 46. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Άρχεται η 47. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία για την 48. Πέρας. Εγκρίνεται. 49. Πόλσεν και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία για τον 49. Πέρας. Εγκρίνεται. 50. Άρχεται η ψηφοφορία για την 50. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Άρχεται η ψηφοφορία για την 51. Ελίζαμπεθ. Εψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται. 52. Άρχεται η ψηφοφορία για την 52. Πέρας. Εγκρίνεται. 53. Πέρας της ψηφοφορίας για την 53. Η 53 μάλλον εγκρίνεται. 5. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβιβαστική 5. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Ψηφίζουμε για την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 60 εγκρίνεται. 61. Άρχεται η ψηφοφορία για την 61. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Άρχεται η ψηφοφορία για την 62. 62 άρχεται ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. 63. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 63. Πέρας, εγκρίνεται. Σε 64. Άρχεται η ψηφοφορία για την 64. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. 66. 66. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας της για την 66. Εγκρίνεται. 67. 67. Άρχεται η ψηφοφορία για την 67. Πέρασε τη ψηφοφορία για την 67. Εγκρίνεται. 68. Τελευταία ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε για την 68. Πέρα. Απορρίπτεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση του συναδέλφου Γκλάτφελντερ. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Ωραία. Με 33 ψήφους υπέρ, 3 κατά και μία αποχή Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και Γκλάτφελντερ. Η Ράσια. Σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη. Μια τελευταία προσπάθεια για να ψηφίσουμε, συνάδελφοι. Σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου Λουίς Μανουέλ Καπόλα Σάντους. Όπως τα ξέρετε, συνάδελφοι, στις 30 Αυγούστου εγκρίναμε 45 τροπολογίες περί προπολογισμού που ε, υποβλήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για το σχέδιο προπολογισμού του 2012. Τώρα πρέπει να περάσουμε σε ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Καπόλα Σάντου για την ε, θέση του Κοινοβουλίου που σε ό,τι το σχέδιο προπολογισμού του 2012, όπω τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο στι 25 Ιουλίου. Συνολικά υποβλήθηκαν 9 τροπολογίε στο σχέδιο έκθεση, αλλά δεν θα δώσω το λόγο στο Λουί γιατί δεν είναι στην αίθουσα. Σωστά. Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε απευθεία. Ξεκινούμε με τον κατάλογο ψηφοφορίας. Είστε έτοιμοι. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε on block. Όχι, όχι γιατί υπάρχουν ε, διαφορές. Ένα. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο. Έναρξη. Άρχεται η ψηφοφορία για το 2, για τη 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τρία. Πέρα. Τρία. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέσσερα. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα. Η τέσσερα εγκρίνεται. Πέντε. ΝΑΤΟ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Πέρας. Η τροπολογία 5 απορρίπτεται. 6. Άρχεται η ψηφοφορία για την 6. Η 6 εγκρίνεται. 7. Άρχεται η ψηφοφορία για την 7. 7. 7. Εγκρίνεται. 8. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία για την 8. 8. Εψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται. Εννέα τέλος. Γέγκλε. Άρχεται η ψηφοφορία για την εννέα. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Τελική ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Τέλεια. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Εγκρίθηκε η θέση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού το 2012 όπως τροποποιήθηκε. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Καπολασάντος. Τζοβάνι, πρόεδρε να ρωτήσω κάτι. προφανώ ετοιμάσαμε έκθεση και στην Επιτροπή Προπολογισμών για το σχέδιο προπολογισμού του 2012. Μια γνωμοδότηση λοιπόν που Ήδη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή αυτή το σχέδιο αποπλογισμού. Νομίζω όμω ότι δεν ήταν τελικά ιδιαίτερα χρήσιμη. Θα πρέπει να οργανώσουμε έτσι το χρονοδιάγραμμά μα, ώστε τα σχέδια γνωμοδότηση να φτάνουν πριν από την ψηφοφορία επί του προπολογισμού, ώστε να έχουν κάποια χρησιμότητα. Με συγχωρείτε. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει να περάσουμε στο σημείο 12. Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες. Η συγγήτρια η Μαρία Νεντέλτσεβα, η οποία είναι ήδη στη θέση της. Συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το θέμα των μόνιμων καλλιεργειών και το σχετικό ντοσχέ, σας ενημερώνω ότι τριμερής διάλογος της 21 Σεπτεμβρίου οδήγησε σε συμβαστική λύση μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κείμενο τη συμβαστική λύση έχει μοιραστεί. Να ευχαριστήσω καταρχήν καταρχάς μάλλον την ομάδα των διαπραγματευτών, ιδίως την κυρία Νεντέλτσοβα για αυτήν τη μεγάλη επιτυχία που κατάφερε να οδηγήσει σε ευτυχές πέρα στην, τον τριμερή διάλογο. Να σου δώσω λοιπόν απευθεία το λόγο Μαρίγια και αν δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνένεση για το θέμα αυτό μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευκόλυνε την σύναψη συμβαστική λύση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θέλω να το πω ευθύ εξ αρχή και να ευχαριστήσω του σκιώδει ηγητέ, καθώ και τη γραμματεία τη Επιτροπή μα, καθώ και του συμβούλου μα που πάσχησαν για να έρθει σε πέρα σε αυτό το θέμα. Στι 31 Σεπτεμβρίου, στον τριμερή διάλογο, καταλήξαμε συμβαστική λύση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και ο συμβασμό αυτό ανταποκρίνεται στου ε, στόχου τη Επιτροπή μα, Επιτροπή Γεωργία. Δηλαδή, θέλουμε αξιόπιστε στατιστικέ, ε, απλουστευμένε και μείωση του διοικητικού άχθου ε, της γραφειοκρατίας και για τις δημόσιες διοικήσεις αλλά και για τους γεωργούς. Στην προπαρασκευαστική συνεδρία για τριμερή διάλογο διαπιστώσαμε ότι υπήρχε συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των πολιτικών ομάδων και συμφωνήσαμε σε ορισμένα θέματα που έπρεπε να θίξουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα τα αναφέρω επιγραμματικά. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα άρθρα 1 και 2 και το παράρτημα, η προτινόμενη διάκριση από το Συμβούλιο που αφορά ε, τις, τα κάτι που ίσχυε για τις ε, μιλιές και τις αχλαδιές, είναι εύλογη, είναι λογικό το θέμα. Τώρα, το βασικό θέμα, το άρθρο 3, η κάλυψη των στατιστικών. Εκεί καταλήξαμε σε βαστική πρόταση που ευθυγραμμίζεται με τις δικές μας τροπολογίες, δηλαδή μείωση του διοικητικού άχθους για τις μικροκαλλιέργειες και για τις εθνικές διοικήσεις. Και τρίτο σημείο, δυνατότητα απόκλησης, εξαίρεσης και ε, διορία που έχουν τα κράτη-μέλη για να τη ζητήσουν. Η εξαίρεση είναι χρονικά περιορισμένη, αλλά περιορίζει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή των συστημάτων τους να προσφύγουν στην αίτηση αυτή για εξαίρεση μέχρι το 2013. Το τελικό κείμενο είναι ικανοποιητικό κατά τη γνώμη μου και κυρίως διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ανταποκρίνεται στους στόχους που είχαμε θεσπίσει από κοινού στην Επιτροπή Γεωργίας. Και πάλι θερμά ευχαριστώ στους συναδέλφους για την προσπάθειά τους, την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ στη Γραμματεία και στους Συμβούλους. Ε, θερμές ευχαριστίες. Μπράβο Μαρία, συγχαρητήρια. Τέλεια. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Αλλιώς έχει εντολή Μαρία να συνεχίσει το καταπληκτικό έργο που ήδη έχει επιτελέσει. Περνάμε στο σημείο 13 που είναι πολύ σημαντικό και πολύ ευαίσθητο. Πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με την μελλοντική ενίσχυση των προβληματικών ζωνών. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας αναγγείλω ότι παρίσταται ο η Γενική Διευθυντρία Λορέτα Μπόρμαν Μαρίνο, που θα μα παρουσιάσει το όραμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική ενίσχυση των προβληματικών ζωνών. Όπω ξέρετε, η Επιτροπή μα είχε λάβει πρόταση από την Επιτροπή πριν την μεταρρύθμιση. Γι' αυτό και είναι σημαντικό στη συζήτηση αυτή να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα τη μελλοντική ενίσχυση. Θα να δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή Μαρίνο και μετά... Κυρία. Την... Κυρία Μαρίνο, συγγνώμη, και ε, Λορέτα Μαρίνο και μετά θα γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ. Για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε τώρα, ε, να σας εξηγήσω ότι ε, ε, μάλλον από πού ξεκινήσαμε και ας θυμηθούμε ποια υπήρξαν τα βασικά βήματα στην διαδικασία εξελίξεως αυτού του θέματος, του φακέλου των προβληματικών ζωνών. Θα αρχίσω με το προήμιο για μια διευκρίνηση η υποστήριξη για τις προβληματικές ζώνες ξεκίνησε το 1975 προβλέποντας τρεις κατηγορίες ορινές, ενδιάμεσες και με συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Θα υπενθυμίσω επίσης τα διάφορα βήματα τα οποία αναφέρονται στις ενδιάμεσες, όχι στις ορινές ούτε σε εκείνες με ειδικά μειονεκτήματα επί των οποίων μέχρι τώρα τίποτε στην ουσία δεν έχει αλλάξει. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στο 2003, οπότε, όταν είχε γίνει μια ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου με βασικό επιχείρημα ότι ήταν ανεπαρκείς οι ενδείξεις που να δείχνουν ότι μπορεί πράγματι να ισχύσει η ταξινόμηση που είχε γίνει των ενδιάμεσων ζωνών και ότι οι χώρες μέλη χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα περίπου 140 ε, δικτών για να καθορίσουν τις ζώνες αυτές. Και στις αρχές ε, της δεκαετίας του 90 υποτίθεται θα γινόταν μια αναθεώρηση. Δεν έγινε όμως λόγω της αντίθεσης ε, ορισμένων χωρών μελών. Το ελεγκτικό συνέδριο τότε είχε συστήσει να γίνει μια σε βάθος επανεξέταση της νομοθεσίας για τις ενδιάμεσες ζώνες και είχε συστήσει επίσης να δημιουργηθεί ένας καταλληλότερος αριθμός δικτών και για τις διάφορες αντισταθμίσεις και για την συνολικότερη αξιολόγηση του προγράμματος. Εν ώψη αυτών των εξελίξεων, στην διάρκεια της ε, φάσεως της προπαρασκευής για την ε, προγραμματική περίοδο 2007 έως 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εργάζεται με την πρόθεση να περάσει από την εθνική οριοθέτηση σε μια κοινοτική οριοθέτηση των ζωνών η οποία να βασίζεται στους δείκτες της παραγωγικότητας όπως για παράδειγμα ε, ο αριθμός των βοσκοτοπιών η, ε, η μέση παραγωγικότητα, η μέση εσοδιά και ούτω καθεξής. Τα οποία να είναι οι δείκτες να είναι διαθέσιμοι ανα πάσα στιγμή σε κοινοτική βάση. Ωστόσο, οι υπολογισμοί, οι μας δείχνουν ότι τέτοια, τέτοιου είδους οριοθέτηση θα οδηγούσε σε μία μείωση των ζωνών κατά 60%. Και αυτό βέβαια βρήκε αντίθετες στις χώρες μέλη. Αυτό λοιπόν που συνέβη τελικά όταν το Συμβούλιο όταν το Συμβούλιο το 2005 ενέκρινε τον κανονισμό 1698 ήταν να διατηρήσει το σύστημα για κάποια περίοδο χρόνου και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα ώστε να υποβάλει προτάσεις για ένα νέο σύστημα οριοθέτησης και πληρωμών από το 2010 και μετά. Επί της ουσίας το Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνταν για την οριοθέτηση και ταξινόμηση των ζωνών και για τους στόχους αυτούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εργάζεται και εργάστηκε από το 2005 έως το 2008 για να εξεύρει, να καταλήξει σε κοινά βιοφυσικά κριτήρια και για να γίνει αυτό το Κοινό Κέντρο Ερευνών ανέλαβε να ε, ορίσει ορισμένα νέα κριτήρια στη βάση του κλίματος και του εδάφους, τα οποία θα αποτελούσαν την βάση μιας απλής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται με συγκρίσιμο τρόπο σε όλες τις χώρες μέλη και που να είναι ανεξάρτητη από τις εσοδίες. Για να γίνει αυτό, ένα πάνελ ε, ε, εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκε και το έργο του ε, συντονίστηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Το, η ομάδα αυτή των ε, εμπειρογνωμόνων κατέληξε σε 8 κριτήρια κλίματος και εδάφους με οριακές τιμές και όπου αυτά έχουν σημαντική επίπτωση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Τα κριτήρια αυτά αξιολογήθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και συζητήθηκαν σε βάθος με τις χώρες μέλη. Και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι οι απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της νέας προσέγγισης οριοθέτησης και οι απαραίτητες κλίμακες ήταν διαθέσιμες ή θα μπορούσαν να συλλεχθούν μόνο στο εθνικό επίπεδο, τα σχετικά δεδομένα δηλαδή. Το έργο αυτό λοιπόν ήταν τόσο δύσκολο και τόσο σε βάθος ώστε η προθεσμία του 2010 που είχε επιβάλει το Συμβούλιο Υπουργών στην Επιτροπή τελικώς δεν έγινε δυνατό να τηρηθεί. Για να μπορέσει το Συμβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, Κοινοβούλιο, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για να μπορέσουν λοιπόν να τηρούνται ενήμερα της διαδικασίας, εξεδώσαμε την ανακοίνωση του 2009 η οποία περιλάμβανε μια ενδεχόμενη νέα ταξινόμηση των ενδιάμεσων ε, ζωνών, πάλι χωρίς τις ορεινές ζώνες και χωρίς τις ε, ζώνες ειδικών μειονεκτημάτων, με 8 βιοφυσικά κριτήρια που έχουν σχέση με το έδαφος και το κλίμα και τα οποία καθιστούν δυνατό να ταξινομηθούν οι ζώνες αυτές με αντικειμενικό, ακριβή, διαφανή και συγκρίσιμο τρόπο. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες των κριτηρίων αυτών, αλλά θα προσθέσω μόνο ότι η ανακοίνωση περιγράφει επίσης τον μηχανισμό που αποκλήθηκε fine tuning και ο οποίος μηχανισμός σε περιπτώσεις όπου οι γεωργοί έχουν κατορθώσει να ξεπεράσουν με επιτυχή τρόπο τους περιορισμούς και να επιτύχουν μια επικερδή γεωργία σε ζώνες με δυσμενείς συνθήκες ο μηχανισμός αυτός ε, θα πρέπει να αφαιρέσει, θα εξυπηρετήσει στο να αφαιρεθούν οι ζώνες αυτές. Έτσι το 2009 το Συμβούλιο ενέκρινε ε, τα σχετικά απορίσματα τα οποία ζητούν από τις χώρες μέλη ε, να κάνουν την αξιολόγηση των βιοφυσικών κριτηρίων και να κάνουν και το fine tuning που σας ανέφερα. Από τότε και μετά Έχει γίνει και τεράστια διμερής προσπάθεια και από τις χώρες μέλη, προσπάθεια λοιπόν στο διμερές επίπεδο, και από τις ε, υπηρεσίες της Κομισιόν που έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να θέσουν υποδοκιμασία τα κριτήρια αυτά. Και οι 27 χώρες μέλη έχουν υποβάλει τα αποτελέσματα των απεικονίσεών τους και έχουν υποβάλει και ε, σε ορισμένες περιπτώσεις και εναλλακτικέ προτάσεις Έχουμε προχωρήσει συζητήσεις μαζί τους σε πολλές διμερείς συναντήσεις, καθώς επίσης και σε συναντήσεις της ε, Επιτροπής Αναπτύξεως της Υπέθρου. Οι συζητήσεις αυτές έχουν καταλήξει σε ορισμένες τροποποιήσεις και προσαρμογές των κριτηρίων. Πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι απεικονίσεις έχουν δώσει ξεκάθαρα στοιχεία ότι η οριοθέτηση στην βάση των βιοφυσικών κριτηρίων είναι διαφανής, είναι συγκρίσιμη και είναι και αξιόπιστη. Επομένως, το θέμα των λιγότερο ευνοημένων περιοχών που συχνά είναι ένα σημαντικό θέμα μπορεί τελικά να στηριχθεί με αντικειμενικά κριτήρια. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα χρονικό σημείο όπου στο μεταξύ ο προβληματισμός για την αναδιάρθρωση της κοινή αγροτικής πολιτικής για μετά το 2013 όχι μόνο έχει αρχίσει αλλά ήδη έχει προχωρήσει πολύ. Είναι λοιπόν φυσικό τα, η νέα οριοθέτηση και τα νέα κριτήρια να ενταχθούν στο συνολικό πακέτο, στη συνολική δέσμη των μέτρων της κοινή αγροτικής πολιτικής για μετά το 2013. Και έχουν λοιπόν ενταχθεί στις προτάσεις που θα απασχολήσουν και θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα και ασφαλώς είμαι διαθέσιμη, διατεθειμένη μάλλον, <clears throat> μετά από την έγκριση από πλευράς της Επιτροπής, να θέσω υπόψη σας όλες τις πτυχές και τις λεπτομέρειες που έχουν περιληφθεί στην πρόταση για την ανάπτυξη της υπαίθρου, την πρόταση κανονισμού για την ανάπτυξη υπαίθρου μετά το 2013. Αυτό που μπορώ να πω για την ώρα είναι ότι η παρούσα οριοθέτηση θα παραμείνει ενισχύει μέχρι τα τέλη του 2013 και <clears throat> θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού τις χώρες μέλη για να επιλύσουμε τα εναπομένοντα προβλήματα και στα επόμενα ένα-δύο χρόνια, ορισμένες χώρες βέβαια περισσότερο, άλλες λιγότερο, θα χρειαστεί να καταβάλουν προσπάθεια για να ε, μας υποβάλουν πιο ολοκληρωμένα δεδομένα καθήκον βέβαια που από την ε, χρηματοδοτική άποψη μπορεί να ενισχυθεί και με τεχνική υποστήριξη ώστε τα νέα αυτά δεδομένα και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν βέβαια νέα δεδομένα αλλά όπου υπάρχουν μπορούν να, η προσπάθεια μπορεί να στηριχθεί από την ε, τεχνική πλευρά από εμάς. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική στήριξη των ζωνών αυτών, στην ανακοίνωσή της του Νοεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ένας από τους κύριους στόχους θα είναι να δίνεται αντιστάθμιση για δυσκολίες παραγωγής σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς για να μην εγκαταλειφθούν οι περιοχές αυτές. Η ανακοίνωση αυτή ορίζει επίσης ότι το, μέλος, το μέλλον μάλλον των πληρωμών αυτών θα βασίζεται στις προσπάθειες ε, διαρκούς και εφόρου αναπτύξεως της γεωργίας σε περιοχές όπου αυτό είναι απαραίτητο με πρόσθετο, πρόσθετη στήριξη εισοδήματο των γεωργών ως συμπλήρωμα στην στήριξη που δίνεται με τον δεύτερο πυλώνα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Και όπως κατανοείτε και εσείς κύριε Πρόεδρε και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση, πριν μια εβδομάδα μόλις πριν από την έγκριση της προτάσεως του νέου κανονισμού να σχολιάσω περαιτέρω σχετικά με το μέλλον των ε, λιγότερο ευνοημένων περιοχών και με αυτά τα λόγια σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Διευθύντρια Μαρτίνο για αυτή την διεξοδική παρουσίαση και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ξεκινάμε με τον κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Διευθύντρια Μαρίνο. Έχω επανειλημμένο ζητήσει να γίνει η συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία. Αυτό που μόλις τώρα μας παρουσιάστηκε επιβεβαιώνει τους ενδιασμούς μου για το όλο θέμα. Η Διευθύντρια μας αφηγήθηκε πώς γεννήθηκε η πρόταση αυτή η οποία την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω αν τυχαία η αποπρόθεση περνάει από το Κοινοβούλιο. Ε, στο Κοινοβούλιο όμως έχουμε εκφραστεί για το όλο ζήτημα και δεν είπαμε αυτά που μόλις ακούσαμε ή από την Διευθύντρια. Δεν τα επαναλαμβάνω, διότι όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά Μιλήσαμε για συνδυασμένα κριτήρια. Είπαμε ότι θα πρέπει η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να διαθετηθεί ως θέμα. Ότι χρειάζεται μεγάλο επίπεδο αλληλεγγύης σε, σε τοπικό επίπεδο. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε μια άλλη πορεία από αυτή που μόλις μας παρουσίασε η Διευθύντρια. Μία ΚΑΠ τελείω διαφορετική, κάτι σαν αυτό που συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιληθεί εφόσον προβλεφθεί κάποια ευελιξία για, τον, για την τρίτη ομάδα των ειδικών περιφερειών. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά επειδή υπήρξε εισηγητή στο Κοινοβούλιο, πρέπει να πω ανοιχτά ότι αισθάνομαι ότι κάπως με, κοροϊδε... με κοροϊδέψανε. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή έχει δύο δυνατότητες. Πρώτον, να ακολουθήσει αυτά που λέει η Επιτροπή, γυρίζοντας την πλάτη σε αυτά που πολιτικός όμως έχει υποστηρίξει το ίδιο το Κοινοβούλιο, ή τουλάχιστον να σεβαστεί τον εαυτό του το Κοινοβούλιο και να συμπεριφερθεί όπως αρμόζει. Πιστεύω ότι για το θέμα αυτό, και θα κλείσω εδώ, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί την ερχόμενη εβδομάδα. Διότι πρόκειται για ένα ζήτημα που ε, πολύ ενδιαφέρει τους γεωργούς. Μην ξεχνάμε ότι με αυτή την πρόταση για πολλά από τα κράτη-μέλη θα αλλάξει ο χαρακτηρισμός ενός τρίτου των ε, προστατευόμενων αυτή τη στιγμή περιοχών. Δεν είναι αμεληταίο και από πολιτική αποψή είναι διατραπέστε το ζήτημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Χέρμπερτ, αλλά προφανώς η πρόταση θα αποτελέσει μέρος του νομοθετικού πακέτου της ΚΑΠ. Θα μας το παρουσιάσει το ή άλλως την επόμενη φορά ο Επίτροπος Τσιόλος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποιο ρόλο θα αναλάβουμε ούτως ή άλλως ε, σε σχέση με αυτό το νομοθετικό πακέτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λάβουμε υπόψη όσα ψήφισε ω τώρα το Κοινοβούλιο και με ευρία πλειοψηφία ε, σε σχέση και με τη δική σου την έκθεση. Ελίζα Μπεθ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενστερνίζομαι απόλυτα αυτά που είπατε. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτά που μας ε, παρουσίασε ο κύριος Ντόρτμαν που εκπώνησε μια πολύ καλή έκθεση. Και δεν νομίζω ότι είναι ο μόνος που αισθάνεται ότι τον έχουν περιπέξει. Και εμείς το ίδιο νιώθουμε έχουμε δικαίωμα εύλογο ε, να ενημερωθούμε για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που δεν συνέβη μέχρι τώρα. Περιμένω λοιπόν από, και από το συνάδελφο Ντόρφμα να συνεργαστεί στενά με τους κοιόδης για να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Γιατί σε ορισμένες χώρες θα πρέπει τα, τα συστήματα να τροποποιηθούν άρδιν και θα γίνουν σφοδρές συζητήσεις σε πολλές χώρες για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απαιτητικοί στη συζήτηση και να γίνει όσο πιο διεξοδικά και εμβριθώς γίνεται. Ο κύριος Στόρτμαν έχει πολύ σαφείς προσδοκίες και απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Μπέθ, Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε ήδη εκτενή συζήτηση για το θέμα αυτό. Το ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάζεται το θέμα από το 2003. Θα ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά και εγώ αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, Ντόρφμαν και Γέγκλε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκυψε με σοβαρότητα στο θέμα αυτό και μάλιστα ο κ. Ντόρφμαν εκπώνησε και σχετική έκθεση που εγκρίθηκε με σημαντική πλειοψηφία και νομίζω ότι η έκθεση αυτή βρήθη πολύ σημαντικών συμβαστικών προτάσεων. Είχαμε και το αίτημα του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε κατά μέρους. Οι συνάδελφοι ζήτησαν να διαφυλαχθεί και να ληφθεί υπόψη ο πυρήνας της έκθεσης Dorfman, κάτι που δεν συνέβη. Υπήρξε μια, ένας κατακαιρματισμός και μια αλλίωση του περιεχομένου. Για να αποκατασταθεί λοιπόν η εμπιστοσύνη μας, θα πρέπει να γίνουν τα εξή βήματα. Να εξεταστεί πρώτα αυτή η έκθεση πέραν της, του πακέτου μεταρρύθμισης ΚΑΠ και να της δοθεί η δέουσα ξεχωριστή θέση που της αξίζει, ώστε να την εξετάσουμε νυφάλια. Κατά τη γνώμη μου θα έχουμε ε, μεγάλη επίβολη μεταρρύθμιση, αλλά το τμήμα που αφορά αυτό το σημείο θα είναι μικρό, ελάχιστο. Και σίγουρα έγιναν πολλά λάθη που ίσως ε, έχουν στην πράξη συγκεκριμένες επιπτώσεις. Εμείς είμαστε πολιτικοί ειδικευμένοι σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Θέλουμε στοχοθετημένες πολιτικές δράσεις. Και όταν διαπράττουμε σφάλματα θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στους γεωργούς για αυτά. Άλλωστε είμαστε και εκπρόσωποι των συμπολιτών μας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Θα πρέπει το θέμα αυτό να περάσει στον Τούκο. Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζω είναι ότι περιοριστήκαμε μόνο στα βιοφυσικά στοιχεία. Παρά είναι περιορισμένη αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι η απερίμωση είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Και ο συνάδελφος Ντόρφαν υπέβαλε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για το θέμα αυτό στην έκθεσή του. Θα παρακαλούσε λοιπόν αυτές οι προτάσεις να ληφθούν υπόψη επικοδομητικά και να μην μπουν σε ένα σιρτάρι και λησμονηθούν, γιατί μια τέτοια στάση πραγματικά είναι εκνευριστική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει συγκεκριμένε αρμοδιότητε. Οπωσδήποτε θα το πράξουμε, κύριε Γιάρ. ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εστερνίζομαι πλήρως ε, αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. δόρφα Γκρέσ ε, και Γιάρ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεντρώσαμε σημαντική πλειοψηφία, διακομματική, για την έκθεση Ντόρφμαν. Και διαπιστώνουμε παρόλα αυτά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη αυτέ τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι υπερβολικό. Νομίζω ότι ε, εμπέζει και περιφρονεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ίδια τη συνθήκη τη Λισαβόνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να τη στείλουμε μερικά αντίτυπα τη συνθήκη τη Λισαβόνα για να ρίξει ματιά. Το δικαίωμά μα που μα δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Η Κομισιόν έχει βεβαίω το δικαίωμα να κάνει προτάσει σχετικά με το πώς θεωρεί ότι είναι τα πράγματα, αλλά την αρμοδιότητα, την αποφασιστική αρμοδιότητα διαθέτουμε εμείς και το Συμβούλιο. Ήταν δε βαρύτατο σφάλμα το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν επεξεργάστηκε το θέμα των μειονεκτικών περιοχών πριν από την μεγάλη μεταρρύθμιση της Γεωργίας. Εγώ είχα ήδη πει ότι οι αποφάσεις αυτές για τις μειονεκτικές περιοχές μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για τη μεγάλη μεταρρύθμιση και δυστυχώς έχασε την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα ρυθμίσει εγκαίρως. Διαπιστώνω και εγώ ότι αυτά τα βιοφυσικά κριτήρια από μόνα τους δεν είναι επαρκή για να κρίνει κανείς ποια περιοχή είναι μειονεκτική και ποια όχι. Και κάτι που δεν βρίσκω σωστό είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει χάρτες για το πώς εφαρμόζονται και μάλλον ποιες επιπτώσεις θα έχει η εφαρμογή των βιοφυσικών κριτηρίων. Θα ήταν πολύ διαφορετικά αν είχαμε τους χάρτες. Από πλευράς της πολιτικής μου ομάδας μπορώ να σας πω καθαρά ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε την ε, συμπεριφορά αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ Άλμπερτ. Μάρτιν Όσλινγκ. Δεν θα βγάλω το ε, ξύφος μου όπως ο ειδικό του Λαϊκού Κόμματος αλλά υπάρχει συνολικά μια εντολή για μια ενοποίηση, ευρωπαϊκή ενοποίηση και στο προκείμενο θέμα και δεν την αρνούμαστε. Τα κριτήρια τα οποία υποβάλλονται τώρα πρέπει να κρίνουμε εάν είναι ικανά, επαρκή δηλαδή, ή αν πρέπει να περιληφθούν και τα κοινωνικο-οικονομικά, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Είναι δύσκολο και είμαι σύμφωνος ότι είναι δύσκολο να γίνει εκ παραλίλου με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και να μεταφέρουμε και προς τα έξω και προς το κοινό, δηλαδή τι θέλουμε στην κοινή αγροτική πολιτική και ταυτόχρονα να κάνουμε και την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών. Κάτι που ασφαλώς θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις περιφέρειες. Βεβαίω και θα υπάρξουν μετακινήσεις ορίων. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι ως τώρα δεν έχουμε στα χέρια μας χάρτες. Εάν προχωρήσαμε σε τελική ψηφοφορία και αν μας ρωτήσουν οι διάφορες οργανώσεις γεωργών κλπ τι απάντηση δίνουμε, θα είμαστε αναγκασμένοι να του πούμε sorry, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Ενώ φαίνεται πως άλλες οργανώσεις έχουν. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πάρα πολύ. Δεν μπορώ λοιπόν να ε, κρίνω και να λάβω αποφάσεις πριν να γνωρίζω τι σημαίνει για την κάθε μια περιφέρεια η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Θα πρέπει να προχωρήσει τώρα η περαιτέρω επεξεργασία με συμμετοχή του Κοινοβουλίου και όχι τόσο πολύ για το αν το χρειαζόμαστε, αλλά πώς θα χειριστούμε το θέμα, σε ποιο ε, χρονικό πλαίσιο, σε ποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά θέλουμε να μας εξασφαλιστεί ότι στο τέλος θα μπορούμε και εμείς να εκφράσουμε άποψη. Ευχαριστούμε Μάρτιν. Ο Τζιμ Νίκολσον. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με πολλοί με τους προλαλήσαντες. Δεν είναι καλή πρόταση αυτή, ούτε η σωστή μεθοδολογία. Και σίγουρα θα έχει ολέθριες συνέπειες, τουλάχιστον στη δική μου περιφέρεια, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που έχει προταθεί. Δεν ξέρω ποιος περιπέζει ποιον εδώ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ε, πώς έχει κατάσταση και από τη στιγμή που είναι δυσαρεστημένος ο εισηγητής να το διαρευνήσουμε. Είναι λάθο να φέρουμε αυτό το θέμα στο επίκεντρο τη μεταρρύθμιση τη ε, κοινή γεωργική πολιτική, γιατί θα χαθεί μέσα στο γενικό τοπίο και θα υποβαθμιστεί αυτό το θέμα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιληφθεί στο θέμα της ανάπτυξης υπαίθρου ίσως. Αλλά να τύχει δέουσας και ιδιαίτερης προσοχής. Και να είμαστε και προσεκτικοί. Μιλούμε για περιοχές που πραγματικά θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση αν αποχαρακτηριστούν το less favorite area από το χαρακτηρισμό αυτό των μειονεκτικών περιοχών και σημαντικό τμήμα του πληθυσμού τους θα εξολοθερευτεί, θα, θα εξαλειφθούν ολόκληρες αγροτικές κοινότητες σας. Μην το ξεχνούμε. Μας λείπουν πολλά στοιχεία, δεν είμαστε αρκετά ενημερωμένοι. Δεν μπορώ να δώσω το πράσινο φως στην πρόταση αυτή. Θα πρέπει να κατατοπιστούμε λεπτομερέστερα. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή, τον κύριο Ντόρφαν. Αναφέρονται πολλά για το έδαφος, για τα βιοφυσικά στοιχεία, για το είδωρ, τους βοσκοτόπους. Θα δούμε τι θα χαρακτηριστεί μειονεκτική περιοχή και τι όχι. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για μας ε, σωστές αυτές οι προτάσεις, ιδιαίτερα και από το πρίσμα της δικής μου περιφέρειας. Κύριε Κόσλιγκερ, ευχαριστώ. Θεωρώ ανεύθυνη την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το σχόλιο του κ. Χόισλινγκ, που χαίρεται για την ενοποίηση της προσέγγισης, εγώ νομίζω ότι αυτό που πλουτίζει την Ευρώπη είναι η πολυμορφία και η ποικιλία και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Και αν εξετάσετε τις περιφέρειες και τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες ε, θίγονται από τα μέτρα αυτά, είναι εκμεταλλεύσεις οι οποίες από μόνες τους δεν μπορούν να σταθούν στην ελεύθερη αγορά. Αλλά κινδυνεύουμε να χάσουμε μεγάλο μέρος αυτής της πολυμορφίας. Πάλι για αυτά τα βιοφυσικά κριτήρια και για τις απεικονίσεις. Ας θυμηθούμε τι προσπάθεια κατεβλήθη στις χώρες μέλη για την δημιουργία των χαρτών αυτών αλλά και για τις απεικονίσεις. Τίθεται το ερώτημα γιατί τα έγγραφα αυτά δεν τα έχουμε μπροστά μας. Γνωρίζουμε, το είπε και ο Τζιμ Νίκολσον, περίπου προς τα που κατευθύνεται η πορεία αυτή και όσον αφορά βεβαίως τις ε, επιπτώσεις της εφαρμογής των βιοφυσικών κριτηρίων. Εμάς μας έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού αναμένω κάποιο σημείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για τις εκμεταλλεύσεις. Εδώ διακυβεύεται και η ίδια η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς θα εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας και στους γεωργούς μας την ε, συμπεριφορά αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τους προλαλήσαντες. Θα θέλαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει τουλάχιστον σε αυτούς που υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις και οι οποίες αγνοήθηκαν και κανείς δεν γνωρίζει για ποιο λόγο. Νομίζω ότι ε, είδαμε μια αυτιστική συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που είναι απαράδεκτο. Αναφέρθηκε και η πρόταση για τα βιοφυσικά κριτήρια που δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις υπεραπόμακρες περιοχές και κυρίως τα υπερπόντια διαμερίσματα που έχουν μια συγκεκριμένη πραγματικότητα του εδάφους που είναι τελείως άσχετη και διαφορετική από αυτή της ε, υπηρετικής Ευρώπης. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τον τριμερή διάλογο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για ορισμένες περιπτώσεις για να υπάρξει πρόοδος χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο και συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ πιστεύω ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε την ομοφωνία του Συμβουλίου για να απορρίψουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο σε αυτό το θέμα μπορούμε να έχουμε ομοφωνία. Ευχαριστούμε, Μισελ. Ρόντουστ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, με συγχωρείτε μια στιγμή να κλείσω το κινητό μου, και εγώ λοιπόν θέλω να καταστήσω σαφές ότι κατανοώ και στηρίζω την δυσαρέσκεια του κυρίου ε, Ντόρφμαν. Και από όσο γνωρίζουμε, θα καταστήσω σαφές τι εννοώ και με ένα παράδειγμα. Όταν ο κύριος Ντόρφμαν έγραψε την έκθεσή του, ρώτησα και εγώ ποια είναι η χαρτογράφηση της περιφέρειάς μου. Και μου έδειξαν μια χαρτογράφηση όπου μια ελώδης περιοχή που έχουμε και που είναι από τις πιο πολύτιμες που έχουμε ε, εμφανίζεται τώρα ως μειονεκτική περιοχή. Εν τω μεταξύ η Ομοσπονδία Γεωργών μας είχε τον χάρτη αυτό και εμείς ως Ευρωβουλευτές δεν έχουμε ούτε ίχνος δει της χαρτογραφήσεως αυτής. Επιτέλους θα ζητήσω να έχουμε επαρκή πληροφόρηση για να μπορούμε να ενημερώσουμε και του ψηφοφόρου μα. Με ρωτούν σε κάθε συγκέντρωση που πηγαίνω τι γίνεται με τις μειονεκτικές περιοχές. Και είμαι υποχρεωμένο να του απαντήσω ότι δεν γνωρίζω. Και αυτό δεν είναι ικανοποιητικό ούτε για μένα ούτε και για τους ενδιαφερομένους. Ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Έκλεισε η συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχει γενικό σύμπνοια μεταξύ μας. Και πάλι έχουμε φτάσει στο γνωστό σημείο. Χθες το συζητήσαμε και με του ε, συντονιστέ τη ομάδα που ήταν παρόντε και στο δείπνο με τον Επίτροπο Σιόλο, ο οποίο ήταν πρόθυμο να ακολουθήσει τι προτροπέ του Κοινοβουλίου. Αλλά σήμερα είχαμε μια πολλωστή απόδειξη από την πλευρά τη Επιτροπή ότι δεν υπάρχει διάθεση να βρεθεί λύση σε σχέση με τι απόψει του Κοινοβουλίου. Θα το πω λοιπόν και στην εκπρόσωπο τη Επιτροπή σήμερα, όπω το είπαμε και χθε το βράδυ τον Επίτροπο Σιόλο. Δεν θα εγκριθεί κανένα νομοθετικό κείμενο γιατί θα, κάνουμε, θα, θα φροντίσουμε να υπερισχύσουν οι δικέ μα νομοθετικέ αρμοδιότητε. Οι αρμοδιότητε που μα αποδίδονται από τη συνθήκη. Σα προσκαλώ λοιπόν να βρείτε έναν τρόπο ώστε το έργο τη Επιτροπή αυτή, οι συζητήσει που γίνονται εδώ, ιδίω όταν υπάρχει ευρία πλειοψηφία, και η οποία διαμορφώνεται μετά από μήνε, εβδομάδε διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ιδάλω κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε θεσμικό πρόβλημα και δεν θα εγκρίνονται πλέον νομοθετικά κείμενα. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διευθύντρια Μαρτίνο, και περνάμε στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Δηλαδή. Βοητσαχόφσκι, θα πρέπει να μας ενημερώσετε ή να αναβάλουμε το σημείο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση και η αποστολή που πραγματοποιήσαμε ε, και τα Κανάρια νησιά είναι πολύ σημαντική αγροτική ζώνη στην Ευρώπη, στην Ισπανία και το ανακαλύψαμε αυτό, γιατί τα Κανάρια νησιά είναι γνωστά περισσότερο για τον τουρισμό στον κόσμο. Σίγουρα είναι σημαντικό ε, τουριστικός προορισμός. Αυτό το διαπιστώσαμε και κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων επαφών που είχαμε. Αλλά διαπιστώσαμε ότι τα Κανάρια νησιά είναι σημαντική και μάλιστα πολύ σημαντική γεωργική περιφέρεια με πολύ σοβαρά προβλήματα και πολλά ακούσαμε γι' αυτά ακούσαμε πόσο δύσκολη είναι η λειτουργία και η εφαρμογή της γεωργίας σε τόσο απόμακρη περιοχή, γιατί είναι πολύ πιο δαπανηρή η καλλιέργεια, είναι πολύ πιο η είναι πολύ πιο υψηλά τα μεταφορικά έξοδα για τα γεωργικά προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρώπη και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός κυρίως στον τομέα της μπανάνας. Με αυτό κυρίως ασχοληθήκαμε. Υφίσταται τα Κανάρια νησιά αθέμητο ανταγωνισμό για τις μπανάνες από τρίτες χώρες και οι οικοδεσπότες μας ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι. Είχαμε πολύ άριθμες συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής κυβέρνησης, της αρμόδιες αρχές. Ήταν πολύ καρποφόρες και επικοδομητικές αυτές οι συναντήσεις και πραγματικά επιστρέψαμε από την αποστολή αυτή πλουσιότερη και πολύ πιο κατατοπισμένη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία σε τόσο απόμακρη περιοχή όπως είναι τα Κανάρια νησιά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη μας από τα Κανάρια νησιά. Τις ευχαριστήσεις τη στείλαμε φυσικά και γραπτός. Πραγματικά ήταν άριστα διοργανωμένη αυτή η επίσκεψη και θερμά ευχαριστίες ε, στον συνάδελφο Μάτο που ήταν πραγματικά η ψυχή αυτής της αποστολής. Ήταν πολύ καλή πρόταση η αποστολή της αντιπροσωπείας μας στους Κανάριες νήσους, γιατί πραγματικά ε, εξοικειωθήκαμε με τα προβλήματα της Γεωργίας σε μια υπεραπόμακρη περιοχή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Βατσαπόσκη. Και μια σημαντική είδηση για τους συναδέλφους για την υποβολή προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει πλέον η προθεσμία. Ε, λίγη στις 11 το πρωί στις 12 του μήνα την ερχόμενη εβδομάδα ώστε να μπορέσει να γίνει συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας ως τις 12.30. Άρα δεν θα υπάρξει συνέντευξη τύπου του Επιτρόπου εφόσον δεν έρθει προηγουμένως το Κοινοβούλιο για να παρουσιάσει τις προτάσεις του. Μετά θα μεταβεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους χώρους της, στα γραφεία της, για να δώσει τη συνέντευξη τύπου. Πρώτα η παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά στους δημοσιογράφους και όχι αντιστρόφως. Σας ε, ενημερώνω ότι χθε με τους συντονιστές πήραμε κάποιες αποφάσεις για ορισμούς εισηγητών και τέλος, πριν σας αφήσω, να σας θυμίσω ότι στις 12 Οκτωβρίου, 11, 12, 12 Οκτωβρίου θα βρεθούμε για αυτήν την σημαντικότατη ημέρα όπου θα γίνει παρουσίαση της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους. Λήξη της συνεδρίασης.